Where ah, Κυρίσω την έναρξη της Συνόδου. Επαναλαμβάνεται η Σύνοδος Ομιλίας που διακόπη τη 7η Απριλίου 2010. Καθίστε σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Proszę Κυρίες και κύριοι, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της 7 η Απριλίου 2010. Έχετε παρατηρήσει από αυτόν, όχι. Θεωρούνται λοιπόν τα πρακτικά εγκεκριμένα. γραπτή δήλωση 71 του 2009 τον λένε ε, Μιχαήλ Τρεμόπουλου, Λίβια Γιαρόκα και Τεότεγκερ για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού και θα διαβεβαστεί αρμοδίως ε, θα συμπεριληφθεί στα κείμενα που θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια της παρούσης συνόδου. Και θα δημοσιευθούν στα αντίστοιχα πρακτικά. Θέλει το λόγο από αυτό η κυρία Λίν. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση που 71 για τον καρκίνο του μαστού. Όπω να ψηφίσετε περισσότεροι, πρόκειται για τον κύριο λόγο θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηλικίε από ηλικίε 35 έω 59 ετών